αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα διαβιβάσω αμέσω, θα θεωρήσω. Λοιπόν, θα στείλω τα δέοντα έγγραφα. Λοιπόν, διακόπτεται η σύνοδος. Καλό σας βράδυ.